Ξεκινήσουμε τη συνεδρίασή μας, αγαπητοί συνάδελφοι. Σας καλωσορίζω όλους. Βλέπω ότι υπάρχουν ε, ορισμένοι βουλευτές που κατάφεραν να έρθουν εν γέρος για τη σημερινή μας συνεδρίαση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. Ας περάσουμε ευθύ αμέσω στο πρώτο σημείο, έγκριση της ημερήσια διάταξη. Υπάρχουν σχόλια, παρατηρήσεις, δεν βλέπω κανέναν. Εγκρίνεται λοιπόν η μερίσια διάταξη, δεν έχω ανακοινώσει, άρα μπορούμε να περάσουμε στο σημείο 3. Απολογισμός της αποστολής των Επιτροπών ΑΦΕΤ και ΣΕΝΤΕ στην Νορβηγία. Έλαβε χώρα η αποστολή αυτή πριν από δύο εβδομάδες. Συνολικά ήμασταν 11 ευρωβουλευτές από την ΑΦΕΤ, Η κύριοι Νταν Πρέντα, Φουντζουλίτσα, η Νίνα Γκίλα, οι κύριοι Καν, Κάρτσκι και Νάρτα και είχαμε και τρεις συναδέλφους από την ΣΕΝΤΕ, Στροντεύσκη, την κυρία Αναγκόμες και τον κύριο Ούρμας Παέτ, καθώς επίσης και τον επικεφαλής αντιπροσωπεία για τη συνεργασία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τι σκανδιναβικέ χώρε συμπεριλαμβανομένε τη Νορβηγία. Είχαμε λοιπόν μαζί μα τον κύριο Γιώνα Ντόρμαν μπορέσαμε μέσω της αποστολής αυτής να εμβαθύνουμε περισσότερο τη σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης και Νορβηγίας, ιδίως τις πολιτικές μας σχέσεις και τις σχέσεις στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας. Είχαμε πολλές υψηλόβαθμες συναντήσεις με τον Υπουργό Εξωτερικών, με τον Υπουργό Άμυνας, καθώς επίσης και με τον Διευθυντή των Μυστικών Υπηρεσιών της Νορβηγίας. Καταφέραμε να εμβαθύνουμε περισσότερο τη γνώση που έχουμε μέσω περαιτέρω διαλόγων και επιτόπου επισκέψεων στην κοινή βάση του ΝΑΤΟ, καθώς επίσης και στην βασική αεροπορική βάση της Νορβηγίας, καθώς επίσης και στο κοινό κέντρο έρευνας και διάσωσης που βρίσκεται στον Πόντο. Είχαμε επίσης επαφές με τους επικεφαλείς του Νορβηγικού Πολικού Ινστιτούτου, καθώς επίσης και με την Ακτοφυλακή και με το Αρκτικό Συμβούλιο στο Τρόμσο και στο Σβάλμπαρνταρ. Επίσης είχαμε επαφή με καθηγητές και φοιτητές από το Πανεπιστήμιο του Σβάλμπαντ, που είναι ουσιαστικά, αν θέλετε, το πιο βόρειο πανεπιστήμιο το οποίο υφίσταται στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον του επικεφαλεί όλων αυτών των οργανισμών από την Νορβηγία, καθώς επίσης και τη δική μα τη γραμματεία για την αποστολή αυτή. Ουδέποτε είχαμε, μπορώ να πω, μια τόσο καλά οργανωμένη αποστολή και επίσκεψη πολύ θετική επίσης και υποδοχή από την νορβηγική πλευρά και ελπίζω ότι πραγματικά θα καταφέρουμε κάποια μέρα και εμείς να ανταποδώσουμε την καταπληκτική αυτή νορβηγική φιλοξενία την οποία δεχτήκαμε. Μέσω της αποστολής αυτής φάνηκε επίσης ότι όχι μόνο αξίζει να πηγαίνουμε στις πρωτεύουσε των χωρών που επισκεπτόμεθα, αλλά μαθαίνουμε πάρα πολλά πράγματα όταν μπορούμε να επισκεφτόμαστε και άλλες πόλεις και άλλες περιοχές. Αυτό είδαμε και στο Σπίνσμπέγκερν, καθώς επίσης και στο Σβάλμπατ, το Μπόντο και τις άλλες περιοχές που επισκεφθήκαμε στην Νορβηγία. Στις 27 Αυγούστου, ημέρα Δευτέρα, εξεδώσαμε και το επίσημο ανακοινωθέν τύπου με τα βασικά συμπεράσματα αυτής της αποστολής. Ολοκληρώνω στο σημείο αυτό και μπορούν τώρα το λόγο να πάρουν και άλλοι συνάδελφοι εφόσον το επιθυμούν. Άννα Γκόμες παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας ότι όντως ήταν εξαιρετική η επίσκεψη αυτή και είναι όντως πάρα πολύ σημαντικό να ευχαριστήσουμε τους, την ορβηγική πλευρά για την πολύ καλή αυτή οργάνωση. Πραγματικά μπορώ να πω ότι ξεπέρασε τις προσδοκίες που είχα η επίσκεψη αυτή, διότι είδα ότι υπάρχει ένα πάρα πολύ σημαντικό δυναμικό βελτίωση και ενίσχυση συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη Νορβηγία, που θα ευχόμουν πραγματικά να ήταν επίσημο μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο βέβαια στην πράξη. Αλλά αυτό το οποίο βλέπουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι υπάρχει μια πολύ ισχυρή συνεργαστία. Χαρήκαμε επίση πάρα πολύ που είδαμε ότι υπάρχουν πολλοί πολιτικοί συνομιλητέ μα στην Νορβηγία που ασχολούνται και αυτοί πάρα πολύ με το Brexit και ανησυχούν πολύ περισσότερο για το Brexit αυτό και δεν μπορούν να καταλάβουν τελικά ποιοι είναι οι βασικοί λόγοι που υποκινούν το Ηνωμένο Βασίλειο στο να πάρει την απόφαση αυτή. Οι ίδιοι οι Νορβηγοί λένε ότι δεν θα πρέπει να συμβεί κάτι τέτοιο, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να ισχύουν συγκεκριμένοι κανόνες, αυτοί που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους οποίους ακολουθεί και η νορβηγική πλευρά, η οποία μπορεί να μην είναι επίσημο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά έχει, όπως σα είπα, πολύ στενές σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι σε πολύ στενή επαφή με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βλέπουν τώρα ότι ε, αν ε, από το Ενωμένο Βασίλειο, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε συνειδητοποιούν ότι πρέπει να καταβάλει κανεί μια τεράστια προσπάθεια προκειμένου να καταφέρει εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση να διατηρήσει στενέ σχέσει με την Ένωση. Μιλήσαμε, όπω είπατε και εσεί, Πρόεδρε, για ζητήματα άμυνα, ασφάλεια. Τα ζητήματα αυτά είναι σημαντικά για του εξή λόγου. Καταρχά ε, είναι άμεσος γείτονα τη Ρωσία η Νορβηγία. Υπάρχει συνεργασία με τη Ρωσία σε πολλού τομεί, όπω για παράδειγμα στην αλληλεία, στην έρευνα και σε άλλου τομεί, Από την άλλη όμω. Η Νορβηγία γνωρίζει πολύ καλά πώ λειτουργεί από πολιτική πλευρά η Ρωσία, πώ συμπεριφέρεται η Ρωσία από πολιτική πλευρά. Θεωρώ λοιπόν ότι ε, είναι ενδιαφέρουσα η δυτή αυτή συνεργασία που έχει η ε, Νορβηγία με τη Ρωσία. Από τη μία πλευρά η Νορβηγία είναι μέρος του ΝΑΤΟ, από την άλλη όμως προσπαθεί να διατηρήσει έναν διάλογο, μια σχέση με τη Ρωσία. Ο άλλος παράγοντας που επηρεάζει και τη δική μας τη δουλειά και τις σχέσεις που έχουμε με τη Ρωσία και κάτι το οποίο είδαμε οι δύο όμως πηγαίνοντας κυρίως στο Σλαμπάτ είναι ότι η κλιματική αλλαγή αντίθετα με αυτό που διατείνονται κάποιοι ανόητοι όντως λαμβάνει χώρα και έχει ήδη μείζονες συνέπειες σημαντικότατες συνέπειες και από στρατηγικής πλευράς και όσον αφορά την άμυνα και την ασφάλεια γιατί ουσιαστικά η κλιματική αλλαγή δημιουργεί νέους διάβλους, νέες οδούς μέσω της ε, Αρκτικής. Και ξέρετε ότι στο μέλλον αυτό μπορεί να σημάνει την ύπαρξη πολλών νέων προκλήσεων και για μας, για τη διατήρηση του περιβάλλοντος, αλλά και πολλές άλλες προκλήσεις ε, πέρα από αυτό ακούσαμε ότι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα είναι αυτό που έχει να κάνει με τον αντίκτυπο της χρήσης πλαστικών, την ρήπαση από πλαστικά και πόσο ουσιαστικά αυτό επηρεάζει όλη την βιολογική αλυσίδα της περιοχής και πώς ήδη βλέπουν τις συνέπειες αυτού του φαινομένου και ήδη προσπαθούν να το καταμετρήσουν από επιστημονικής πλευράς μέσω των διαφόρων ερευνητικών Ινστιτούτων που έχουν στην περιοχή. Ήταν επίσης πολύ ενδιαφέρον να δούμε ποια συνεργασία λαμβάνει αυτή τη στιγμή η χώρα με την Ρωσία, αλλά ακόμα και με την Κίνα. Στο Σλαμπάντ πάλι το είδαμε αυτό. Μας είπαν ότι ήδη στο Σβάλμπαρντ ε, έχουν παρουσία οι Κινέζοι, κυρίως ε, για επιστημονικά ζητήματα τα οποία βέβαια ενδιαφέρουν ιδιαίτερα και την Κίνα και τη Ρωσία και όλους τους υπόλοιπους που είναι παρόντες στην περιοχή. Ξέρουμε όμω ότι η επιστημονική έρευνα μπορεί να καλύψει πάρα πολλού τομεί πέρα από την καθαρή επιστήμη και ξέρουμε τι επιπτώσει μπορεί να έχει η τήξη των πάγων στην περιοχή του αρκτικού κύκλου. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν, περισσότερο από ποτέ, να δούμε τη σχέση έχει αυτή τη στιγμή η Νορβηγία ή τι διάλογο αυτή τη στιγμή προωθεί η Νορβηγία με χώρες όπως η Ρωσία και η Κίνα. Και αυτός είναι ένας ακόμα λόγος που πρέπει εμείς να δώσουμε την απαραίτητη προσοχή, τη δέουσα σημασία στις σχέσεις μας με την Νορβηγία. Πήγαμε επίσης ε, σε αυτό το καταπληκτικό επίγειο δορυφορικό κέντρο που βρίσκεται στο Σφάλμπαρντ, όπου ξέρετε ότι ε, Υπάρχουν εκεί πέρα δέκτες που λαμβάνουν πάρα πολλές πληροφορίες από τους ε, δορυφόρους και τις οποίες διαχέουν έπειτα προς διάφορους ευρωπαϊκούς οργανισμούς όπως η ΕΜΣΑ ή προς διάφορες ιδιωτικές εταιρείες. Είναι απίστευτο πραγματικά θα έλεγα να βλέπει κανείς το κέντρο αυτό και να συνειδητοποιεί τελικά πόσα δεδομένα διαχέονται στον υπόλοιπο κόσμο και είναι ασύλληπτο να συνειδητοποιεί κανείς τελικά πόσες επενδύσεις έχουν γίνει από τις νορβηγικές αρχές και από τον ιδιωτικό τομέα στο κέντρο αυτό. Και όντω υπάρχουν πολλοί οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ΕΝΙΣΑ, η ΕΣΑ, η ΕΜΣΑ, οι οποίες συνεργάζονται με το δορυφορικό αυτό κέντρο. Και είδαμε επίσης ότι υπάρχει και ένα τεράστιο δυναμικό περαιτέρω βελτίωσης τη που μπορούμε να έχουμε με το κέντρο αυτό, συνεργασία που ξεπερνά τι καθαρά επιστημονικέ εφαρμογέ. Πρόεδρο, σα ευχαριστούμε, Αναγκόμε, για τι παρατηρήσει αυτέ. Υπάρχουν άλλοι συνάδελφοι που θα ήθελαν να πάρουν το λόγο, να προσθέσουν κάτι σε αυτή τη φάση. Δεν βλέπω κανέναν. Για άλλη μια φορά, λοιπόν, Ολοκληρώνοντα με το σημείο αυτό, πρέπει να πω ότι ήταν εξαιρετική αποστολή αυτή. Πραγματικά υπήρχε μία καταπληκτική προστιθέμενη αξία και νομίζω ότι θα πρέπει να συνεργαζόμαστε όλο και περισσότερο με τους συναδέλφους από την νορβηγική πλευρά και αναφέρομαι τόσο σε εκπροσώπους του Νορβηγικού Κοινοβουλίου όσο και στου εκπροσώπους της εκάστοτε Νορβηγική κυβέρνησης. Ας περάσουμε τώρα στο σημείο 4 της ημερήσια διάταξης και επομένω ε, θα μελετήσουμε ως Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων την ενδιάμεση έκθεση για το πολιτε δημοσιονομικο δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027. Ε, η έκθεση αυτή θα αποτελέσει την πρώτη επίσημη εντύπωση του Κοινοβουλίου στην πρόταση που έκανε η Κομισιόν τη Δευτέρα Μαΐου. Ε, η συμβολή μας ακολουθεί και ήδη εκπεφρασμένε θέσει, όπω α πούμε η θέση που έχουμε εκφράσει όσον αφορά την υλοποίηση των εξωτερικών χρηματοδοτικών εργαλείων ε, του Ιανουαρίου. Ε, η συγγητριά μας είναι η κυρία Μαρίτια Σάκε, η οποία δυστυχώς δεν μπορεί να είναι σήμερα εδώ. Ε, και επομένως μου ζητήθηκε από την Άλντε να διαβαστεί η δήλωσή της. Είναι κάποιος από την Άλντε? Λοιπόν, θα διαβάσω εγώ επομένως τη δήλωση της Μαρίτσιε. δήλωση τη ε, εισηγητρία Μαρίκη Χάκη, εισηγητρία για το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο, λαμβάνοντα υπόψη ε, τι συνολικέ προκλήσει ε, ε τι οποίε αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει αρκετή χρηματοδότηση για όλε τι πολιτικέ Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, Ταυτοχρόνω, ε, η αρχιτεκτονική ε, διαμοιρασμού αυτών των κονδυλίων θα πρέπει να ανταποκρίνεται στα αρχικά μα κριτήρια, που και αυτά με τη σειρά του θα πρέπει να ανταποκρίνονται στι αρχέ και τι αξίε μα. Η Κομισιόν δεν είχε κάνει συγκεκριμένε προτάσει όσον αφορά ε, την μελλοντική δομή διακυβέρνηση ε, μέσω τη οποία ε, θα προωθηθεί ε, ή θα προωθηθεί η χρηματοδότηση. Αυτό θα μπορούσε ε, να ε, δυναμητήσει την θέση της Ευρωπαϊκής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά τις μελλοντικές διαπραγματεύσεις. Θα πρέπει να είμαστε σε πλήρη διαφάνεια. Σωστοί μηχανισμοί και επιτήρησης αλλά και διαφάνειας είναι απαραίτητα έτσι ώστε να γίνει πιο αποτελεσματική χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως επικεφαλής της ομάδας για το εξωτερικό χρηματοδοτικό εργαλείο. Προσδοκώ καλύτερη συνεργασία όσον αφορά ε, τα συγκεκριμένα θέματα τα οποία περιέχονται στο πολιτές δημοσιονομικό ε, πλαίσιο και ε, αναφέρονται ακριβώς στο εξωτερικό χρηματοδοτικό εργαλείο. Αυτά ήθελε να μας πει η συγγήτρια κυρία Μαρίτια Σάκε. Και τώρα θα δώσω το λόγο στα άλλα μέλη της ε, Επιτροπής μας, έτσι όπως καταγράφονται στον κατάλογο των αγοριτών. Αλλά φαίνεται ότι κανείς δεν έχει ζητήσει να εγγραφεί στον κατάλογο των αγοριτών και επομένως... Ε, Στρέφαμε προς τους συναδέλφους, μήπως κάποιος έχει αλλάξει γνώμη, μήπως κάποιος από τους συναδέλφους θέλει να πάρει το λόγο. Ο κύριος Παντζέρη, παρακαλώ. Πρέγκο, λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα φυσικά να ευχαριστήσω ε, και ε, την κυρία Σάκη και σας που διαβάσατε το υπόμνημά της. Ε, δύο-τρία σημεία θέλω να καταγραφούν στα πρακτικά. Πρώτα απ' όλα, κατά τη δική μας άποψη, θα πρέπει οπωσδήποτε να κατανοηθούν σωστά ε, τα, ε, ε, τα κονδύλια τα οποία αφορούν την εξωτερική πολιτική, διότι η κοινή εξωτερική πολιτική είναι εκ των ουκάνευ προϋποθέσεων για την Ευρωπαϊκή Ένωση και επομένως, ναι, θα πρέπει να, υπάρχουν, να υπάρχει χρηματοδότηση των χρηματοδοτικών εργαλείων, αλλά με σωστή παρακολούθηση. Η ίδια η συγγήτρια ε, ε, είναι επικεφαλής της ε, ομάδας που ασχολείται με τα εργαλεία αυτά, αλλά δεν έχει εντολή ελέγχου. Δεύτερον, πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία, η οποία θα επιτρέψει τη μόχλευση επιπλέον πόρων. Τέλος, όσον αφορά τα καταπιστεύματα, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή όλων ε, στο γεγονός ότι ε, τα 10 και μισό δις ε, της, του Ταμείου για την ειρήνη, έτσι όπως το πρόθεσε η Φεντερίκα Μογερίνη το προηγούμενο Ιούνιο, στην ουσία ασχολείται κυρίως με διαδικασίες και ασχολίες ασφάλειας και και ε, άμυνας ε, και επομένως νομίζω ότι θα πρέπει να το μετονομάσουμε σε εργαλείο για την υποστήριξη της ειρήνης. Ε, οπωσδήποτε και όλα τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να τίθενται υπό τον έλεγχο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Παντζέρη, λέει ο Πρόεδρος. Μήπως κάποιος άλλος θέλει να πάρει το λόγο. Η κυρία Λόζινγκ sah und sprach. Bitte. Εκτός μικροφώνου, κυρία Λόιζινγκ. Ναι. Η κυρία Σχάκια δεν είναι εδώ. Και φυσικά παρακολουθώ τη συνεδρίαση από τον υπολογιστή. Να την ευχαριστήσω εκ βάθους καρδίας για την γνωμοδότησή της και σε μεγάλο βαθμό την υποστηρίζουμε. ιδιαίτερως σε ό,τι αναφέρει το 2 της χρηματοδότησης για ό,τι αφορά τη διατήρηση του εργαλείου γειτονία και του Έλλη. Και στο σημείο 3 και 4 συμφωνούμε. Ωστόσο, θα καταθέσουμε τροπολογίες σε ό,τι αφορά το αναπαρατρίο, το δικαίωμα για κοινοβουλευτικό έλεγχο. Θέλουμε να το τονίσουμε αυτό. Το τελευταίο σημείο δεν το υποστηρίζουμε, δεν προκαλεί έκπληξη αυτό, γιατί θεωρούμε ότι δεν είναι νόμιμο να χρηματοδοτούνται στρατιωτικοί εξοπλισμοί από τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρο. Άλλο κανεί που θα θέλει να πάρει το λόγο. Μάλιστα, να δώσω λοιπόν το λόγο στον κύριο Φέλεξ Φερνάνδε Σου. Ξέρω ότι είστε εδώ, αλλά πού κάθεστε. Άννα, εκεί. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω κι εγώ, γιατί σήμερα μπήκαμε στο Κοινοβούλιο χωρίς έλεγχο. Πρώτη φορά πρωτόγνωρο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και νομίζω ότι το ίδιο ισχύει και για τους ε, εκπροσώπου του Κοινοβουλίου που έρχονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νομίζω ότι αυτό διευκολύνει την ζωή μα. Σε ό,τι αφορά την έκθεση τη κυρία Χάκη, να κάνω κάποια σχόλια. Καταρχά να ευχαριστήσω για την συνεκτική προσέγγιση, να ευχαριστήσω για την υποστήριξη, για την αύξηση των κονδυλίων. Πολύ σημαντικό από πλευρά της Επιτροπής σας και προφανώς θα θέλουμε να διατηρηθεί το στοιχείο αυτό, γιατί υπολογίζουμε σε νέα κονδυλία. Καθώς ε, θα συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις ε, για τα κονδύλια, θα, γίνει, θα υπάρξει μεγάλη πίεση σε ό,τι αφορά τα πόσα για την εξωτερική πολιτική. Χρειαζόμαστε μια φιλόδοξη ατζέντα και άρα θα πρέπει να υπάρχουν τα πόσα αυτά. Δεύτερο στοιχείο που θα ήθελα να τονίσω, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης για την Υποσαχάριο ε, Αφρική, για την Κρεβική, τον Ειρηνικό, προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μπουν στον προπολογισμό. Αυτό θεωρώ ότι από μόνο του ενισχύει την ε, παρουσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην εξωτερική πολιτική και μέτρα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που ελήφθησαν για παράδειγμα πρόσφατα δεν θα μπορούσαν να έχουν ληφθεί χωρίς το Κοινοβούλιο αν είχε μπει στην προπολογισμό η αναπτυξιακή βοήθεια σε ό,τι αφορά τώρα τη δομή. Συμφωνώ με αυτά που διαβάσατε. Θα πρέπει να υπάρχει μια ενίσχυση της πολιτικής μέσω της δομής και να προωθηθεί και η πολιτική εποπτεία από πλευρά του Κοινοβουλίου για τις αποφάσεις που λαμβάνονται στο εξωτερικό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό λοιπόν που καλούμαστε θα θέλαμε μάλλον να τονίσουμε σήμερα ότι και από την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης αλλά και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνουμε ένα ενιαίο εργαλείο, να υπάρχει μία ενιαία πολιτική. Σε ό,τι αφορά τα θέματα γειτονίας, ανθρωπινών δικαιωμάτων, θέλουμε όλα αυτά να υπαρχούν στο ίδιο εργαλείο, προκειμένου να υπάρχει και μεγαλύτερη ευελιξία και μεγαλύτερος αντίκτυπος από τη βοήθειά μας. Η πρόταση επίσης ενισχύει το πλαίσιο ενίσχυσης και εποπτείας και την ευελιξία του και την προβλεψιμότητά του και επιμένουμε ότι η ευελιξία δεν εμποδίζει την επιτεύξη των στόχων μας σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, το οποίο άλλωστε και η κυρία Σχάκε το αναφέρει στο σχέδιο γνωμοδότησης. Για τα θέματα άμυνας δεν θα σχολιάσω, δεν είναι ο ρόλος μου άλλωστε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Κύριε Φερνάνδες, από τη Γενική Διεύθυνση ΤΕΦΚΟ, σας ευχαριστούμε. Και τώρα, ο Φιλιππέτρο Τσεριάν Τζεμπριγκόντι είναι εδώ. Εδώ είστε. Έχετε το λόγο από την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και ναι, να συμπληρώσω και εγώ από πλευρά μου αυτά που είπε ο συνάδελφο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να τονίσω κάποια στοιχεία. Καταρχά, καλώ ορίζουμε το σχέδιο τη γνωμοδότηση από πλευρά τη Επιτροπή σας και θα ήθελα να σχολιάσω επίση το σημείο 3 για τη διατήρηση των στόχων της ε, πολιτικής γειτονία και του εργαλείου για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πιστεύουμε ότι οι προτάσει της Ευρωπαϊκή Επιτροπή. ακριβώς προς την κατεύθυνση αυτή κινούνται τα κονδύλια για την πολιτική γειτονία, τα κονδύλια για το εργαλείο ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοκρατίας μπαίνουν μέσα στο εργαλείο αυτό και αυξάνονται κατά 24 και 15% αντιστοίχως και οι συγκεκριμένες ε, ρήτρε του εργαλείου όπως έχουν σήμερα, διατηρούνται ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το μηχανισμό για την ε, γειτονία, για την ε, προγραμματισμό και την ε, εκχώρηση πόρων και στο άλλο εργαλείο ε, σε ό,τι αφορά τις δράσεις απουσία κυβέρνησης και για την χρηματοδότηση μη καταχωρισμένων οντοτήτων, όπως για παράδειγμα οι ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ένα άλλο θέμα για την ε, διαχείριση των εργαλείων. Η κυρία και καλεί να αναπτυχθούν τρόποι για να υπάρχει υποπτή από πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πιστεύουμε ότι αυτό το ενιαίο εργαλείο θα επιτρέψει τη διεξαγωγή ευρύτερου διαλόγου μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Κοινοβουλίου σε πολιτικό επίπεδο. Και θα βρούμε νέους τρόπους ε, διεξαγωγής του διαλόγου αυτού. Άλλα δύο ίσονος σημασίας σημεία. Αν υπάρχει ανησυχία ότι του εργαλείου ανάπτυξης γειτονία για την ασφάλεια και την ε, μετανάστευση θα μπορούσαν ενδεχομένω οι πόροι να μην ακολουθήσουν τους στόχους που έχουν τεθεί. Πιστεύω ότι το θέμα της μετανάστευσης και της ασφάλειας είναι επικαιρό όταν μιλάμε για τις σχέσεις και την εταιρική σχέση που έχουμε τις χώρες αυτές. Ιδάλλως έχουμε άλλα ξεχωριστά εργαλεία για τη μετανάστευση και την ασφάλεια. Έχουμε εσωτερικά κεφάλαια στον προπολογισμό, το ενισχυμένο εργαλείο για τη μετανάστευση. Έχουμε επίσης και την πρόταση στον ε, εξωτερικό κλάδο να δημιουργηθεί μια νέα σχετική ευρωπαϊκή διευκόλυνση. Σε ό,τι αφορά τα σχόλια του κ. Παντσέρη, λοιπόν, θα ήθελα να πω ότι η ενίσχυση των Αφρικάνων εταίρων προκειμένου να μπορούν να διαδραματίζουν ρόλο ειρηνοποιού στην επικράτεια τους αποτελεί έναν τρόπο πρόθεσης της ειρηνής. Και βοηθά στη διατήρηση της ασφάλειας με συνολικό τρόπο, με ενιαίο τρόπο. Πιστεύουμε λοιπόν ότι υποστηρίζουμε τελικά την ασφάλεια και την ειρήνη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θέλει να πάρει κανείς άλλο το λόγο. Δεν νομίζω. Επομένως, η προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών είναι η 18η Σεπτεμβρίου, 11 η ώρα το πρωί. Δηλαδή, έχετε μία μέρα παραπάνω από ό,τι προβλεπόταν αρχικά. Κατά πάσα πιθανότητα θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή μας 8 ή 9 Οκτωβρίου. στην καθήλυνη Ηρμόδια Επιτροπή Προπολογισμών θα ψηφίσουν στις 5 Νοεμβρίου και το ζήτημα αυτό θα περάσει στην πρώτη Ολομέλεια του Νοεμβρίου. Πολύ ωραία. Δεν βλέπω παρατηρήσεις από τη δική σας την πλευρά. Η κυρία Πατρίτσια Φλόρ φτάνει τώρα εδώ πέρα στην αίθουσα. Είναι καθοδόν. Πολύ ωραία. Δεν μπορούμε προφανώ να περάσουμε στο επόμενο σημείο τη μερική διάταξη αν δεν έχουμε μαζί μα την κυρία Φλόρ. Είναι πάντω καθοδόν. Σα προτείνω να κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα μέχρι να φτάσει. Δεν νομίζω ότι θα κάνει πολλή ώρα, επομένω το καλύτερο είναι να μείνουμε στην αίθουσα. Ευχαριστώ.